τομέα των οποροκυπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά, κύριε Σίτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε. Είναι προχωρημένη η ώρα, γι' αυτό θα είμαι λακωνικός όπως το απαιτούν και οι περιστάσεις. Είναι πολύ σημαντική έκθεση γιατί επηρεάζει πολλούς γνωστούς γνωστέ οργανώσει παραγών και ενώσει οργανώσεων παραγών στα κράτη-μέλη. Είναι διαφορετικό το επίπεδο οργάνωση, κάτι που δείχνει το διαφορετικό σημείο αφετηρία των οργανώσεων αυτών στα διάφορα κράτη-μέλη. Μερικές φορές όμως οφείλεται η χαμηλή οργάνωση και στην αποτυχία μια των πολιτικών. Γι' αυτό και θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην οργάνωση των παραγωγών σε οργανώσει, ιδιαίτερα στα προκυπευτικά. Μία μελέτη του Πανεπιστημίου Βάνιγκεν Φυσικά την προσοχή μας στην έλλειψη ασφάλειας δικαίου, κάτι που είναι σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη οργανώσεων παραγωγών και θα ήθελα να παρακαλέσω τον Επίτροπο να απλουστεύσει τις αντίστοιχες διατάξεις για τα απορροκυπευτικά. Επίσης, ε, θα πρέπει να προβλεφθούν κονδύλια για να ε, δούμε το θέμα της διαχείρισης και την άμεση επαφή των οργανώσεων παραγωγών με τους παραγωγούς γιατί ε, μπορεί ένα παραγό να είναι ικανό, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι καλό διαχειριστή. Θα πρέπει λοιπόν ε, να μπορούν οι οργανώσει παραγών να προσλαμβάνουν διαχειριστέ ε, και αυτό είναι σημαντική καινοτομία και που περιλαμβάνει η έκθεσή μου. Επίσης, τα μέσα πρόληψης και διαχείριση των κρίσεων δυστυχώς δεν χρησιμοποιούνται και δεν αξιοποιούνται δεόντως. Γιατί οι κρίσεις δεν οφείλονται μόνο στις διάφορες καταστάσεις αγοράς, μπορεί να οφείλονται σε υγειονομικούς παράγοντες, ακόμη και σε πολιτικούς παράγοντες όπως ήταν το πρόσφατο ρωσικό εμπάργο. Γνωρίζουμε ότι ε, η αγρότες μας βρέθηκαν εκτεθειμένοι ε, στην πολιτική αυτή κρίση με τη Ρωσία και υφίστανται τα αρνητικά αποτελέσματα του ρωσικού εμπάργου. Από την έκθεσή μου ζητάω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της και να προστατεύσει τους παραγωγούς κυρίως από τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, ιδιαίτερα των μεγάλων αλυσίδων διανομής και των μεγάλων λιανεμπόρων που επιβάλλουν ε, τιμές ε, ε, τόσο χαμηλές και ξεφτυλιστικές που συντρίβουν ουσιαστικά τους παραγωγούς. Ένα από τα προβλήματα ε, στην οποία στα οποία πέστησα την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η ανάγκη να εξασφαλιστεί η, ε, η διόνυση της γεωργίας να δίνεται η σκητάλη από γενιά σε γενιά. Να μην σταματάει η γεωργία σε μία γενιά και να υπάρχει ανανέωση. Επίσης, 7,5% μόνο των γεωργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτω των 35 ετών. Αν έχουμε πιο ελκυστικές και πιο αποτελεσματικές οργανώσεις παραγωγών, πολύ περισσότεροι νέοι θα βρουν στη γεωργία εναλλακτική επαγγελματική διέξοδο. Αυτά, επειδή έχουμε φτάσει ήδη κοντά στα μεσάνυχτα, θα είμαι σύντομος. Ελπίζω αύριο το πρωί να υπερψηφιστεί έκθεση. Θα εκφράσω και εκεί κάποιες απόψεις για να μην μακρηγορήσω σήμερα. Σας ευχαριστούμε κύριε Μέλλο για την επίοικιά σας. Έξι συναδελφοί ζήτησαν το λόγο για τη διαδικασία κατσιδιά. Η πρώτα η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να συγχαρώ τον εισηγητή μας κύριο Νονομέλο για την πολύ αξιόλογη έκθεσή του πιστεύω ότι θα πρέπει να απλουστεύσουμε και τις ευρωπαϊκές αλλά και τις εθνικές διαδικασίες για την ε, ίδρυση και καταχώρηση των οργανώσεων παραγωγών και να ελαφρύνουμε το γραφειοκρατικό τους άχθος. Επίσης θα πρέπει να στηρίξουμε ε, τους, ε, παραγωγών ε, σε όλα τα επίπεδα και να δώσουμε κίνητρα για την ίδρυση τέτοιων οργανώσεων παραγωγών προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και το γεωργικό εισόδημα, κάτι που δεν ισχύει μέχρι στιγμή. Είναι χαμηλό το επίπεδο οργάνωση ε, σε οργανώσει παραγωγών και κυρίω η μικρή παραγωγή απορροκυπευτικών αποκλείονται από τέτοιε οργανώσει. Ε, γι' αυτό και χάνουν τα άμεσα ωφέλη του ευρωπαϊκού συστήματο τέτοιοι μικροπαραγωγοί, ενώ η εισαγωγή φρούτων και λαχανικών αυξάνεται και οι ντόπια παραγωγή εκτίθενται σε αθέμητο ανταγωνισμό και αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ. Είναι υπερβολικά περίπλοκη διαδικασία, ιδιαίτερα στην Κροατία και γι' αυτό ζητώ από το Υπουργείο Γεωργία να θεσπίσει εθνικά προγράμματα για να εξασφαλίσει καλύτερη συμμετοχή ε, των ε, Κροατών Γεωργών στο νέο Καθεστώ. Ευχαριστώ κύριο Φραντσουλίτσα για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε τη θέση των οργανώσεων των παραγωγών όσον αφορά την αλυσίδα για να του δώσουμε και κάποιο είδου κίνητρα για αυτέ τι ενώσει των παραγωγών και να υπάρχει διεθνή συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τι ενισχύσουμε αυτέ τι οργανώσει παραγωγών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη γεωργική πολιτική. Θα πρέπει εμένα να υπάρξει ενθάρρυνση σε όλα τα επίπεδα, ιδίω στα κράτη-μέλη που έχουν κάποιε οργανώσει που δεν είναι τόσο πολυάριθμε. Πιστεύω ότι οι οργανώσει παραγωγών μπορούν να βοηθήσουν ε, ε, να λειτουργεί καλύτερα η, η αλυσίδα εφοδιασμού και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όλοι αυτοί οι παραγωγοί έχουν ε, ε, φυγεί από την ρωσική απαγόρευση η οποία θα επεκταθεί το 2016 να συνεχίσουμε με μέτρα στήριξης ε, μέχρι ότου η αγορά επανέλθει στο φυσιολογικά. Αλλά θα πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε να επιβάλλουμε μέτρα βάρος των Ρώσων. Κύριος Μαριάς. κυρία πρόεδρε οι έλληνες παραγωγοί οπωροκυπευτικών προϊόντων παρότι έχουν υποστεί τεράστια ζημιά από το ρωσικό εμπάργκο εντούτοις πήραν ψίχουλα ως αποζημίωση. επίσης οι φτωχοποιημένοι από το μνημόνιο έλληνες παραγωγοί οπωροκυπευτικών έχουν υποστεί φέτος τεράστια ζημιά στην παραγωγή τους και λόγω των θεομηνιών που έπληξαν την πατρίδα μου. ταυτόχρονα συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης των μεγαλοεμπόρων η τρόικα με τις προτάσεις της διαλύει τον πρωτογενή τομέα στην ελλάδα και ζητά την κατάργηση πρώτον των ειδικών καθεστώτων για τους αγρότες και δεύτερον των επιστροφών στο πετρέλαιο κίνησης ενώ προωθεί την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης των κερδών των αγροτών. και όλα αυτά παρότι το εισόδημα των ελλήνων αγροτών μειώθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ και οι φόροι που κατέβαλαν αυξήθηκαν κατά. 150% θα πρέπει λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη στήριξη στον τομέα των οπωροκυπευτικών στην ελλάδα καθώς χωρίς την ενίσχυση αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολο να στηριχθούν και να προχωρήσουν οι νέοι παραγωγοί οπωροκυπευτικών προϊόντων. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο στοιχεία που τα αναφέρετε στην έκθεσή σας και που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλή. Ε, αναφέρατε τη φιλοδοξία σας της αναβάθμισης της ποιότητας και ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει με αυτό το σημαντικό της ατού, της ποιότητας των προϊόντων της, των φρούτων και λαχανικών της. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο η ποιότητα και η αυθεντικότητα, η γνησιότητα είναι πολύ σημαντική, γιατί έχουμε προστατευμένα προϊόντα και στα φρούτα και λαχανικά προστασία της ε, προέλευσης είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό ατού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ποιότητα και η γνησιότητα, η αυθεντικότητα. Δεύτερο σημαντικό θέμα που αναφέρεται είναι οι νέοι. Πολύ αξιόλογοι οι τους νέους στη γεωργία. Νομίζω αυτή είναι πολύ σημαντική ανάγκη, επιτακτική μας ανάγκη για να έχουμε ανανέωση της γεωργίας μας και να έχει και η γεωργία λαμπρό μέλλον και να διονυστεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιέγκας. Η κατάσταση είναι παράδοξη. Έχουμε μια περίμωση των γεωργικών ε, περιοχών, κυρίως ε, των, ε, περιοχών που παράγουν φρούτα και λαχανικά, αλλά έχουμε και μία της κατανάλωσης ε, χαμηλότερο και από τις ε, ε, προτάσεις της ΠΟΗ. Ενώ έχουμε ταυτόχρονα τις μεγάλες βιομηχανίες που εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Θέλουμε μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των οργανώσεων παραγωγών, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Ταυτόχρονα χρειάζονται περισσότερα μέτρα στήριξης και διεύρυνση των και ενίσχυση των δαπανών προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την επιβίωση αυτών των οργανώσεων παραγωγών. Ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους, ε, τις οργανώσεις παραγωγών να αντιμετωπίσουν τις απειλές του τομέα, που είναι κυρίως η υπεροχή των μεγάλων αγρισίδων διανομής. Επίσης, ε, θα πρέπει να, ε, να σταματήσουμε την τάση φιλελευθεροποίησης της ΚΑΠ, που τίποτα καλό δεν θα επιφέρει στη γεωργία μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαστιά. Σεμπαστιά, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια κύριε Μέλλο για το, την άρεστη εκθέσή σας. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση και ξεκαθαρίζει ποια είναι τα βασικά προβλήματα όσον αφορά τα προγυπευτικά. Πρώτα-πρώτα έχουμε αθέμη τον εγωνισμό από τις τρίτες χώρες γιατί παράγουν με κοινωνικές προϋποθέσεις και περιβαλλοντικές που εδώ απαγορεύονται. Έχουμε επίσης τις μεγάλες αλυσίδες που πληρώνουν πάρα πολύ ως τους παρόγους και μιλάμε τώρα για κάποιον κλάδο που κυρίως ε, υπάρχει στην Νότιο Ευρώπη και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα οπότε θα πρέπει να ληφθούν μέτρα επιγόντως αλλιώς πρόκειται να καταληφθεί η ύπεθρος υπάρχει αστιφιλία από τους νέους ε, ε, αισθάνονται προδομένοι, καταλημμένοι από την Ευρώπη οι καλλιεργητές των ότι έχουν δίκιο και στην Βαλένθια την πόλη μου είδα οι συνεταιρισμοί ε, πόσο καλά δουλεύουν. Θα πρέπει επομένως αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν κατεπηγόντως. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος. Ευχαριστώ. Τελευταίος κύριος Χολτ. Σε ευχαριστώ. Δεν θα μείνω στα θέματα της ΚΑΠ εν γέννη. στο UKIP είμαστε και ξέρουμε ότι αυτά καλύτερα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Αλλά θέλω να σας αναφέρω τρία άλλα θέματα που έχουν σχέση με την έκθεση. Πρώτα-πρώτα μπράβο στον εισηγητή γιατί λέει ότι το, απλό είναι σοφότερο και άρα και το πιο απλό σύστημα είναι το πιο καλό για του ε, καλλιεργητές. Συμφωνώ επίση. ότι είδαμε οι νέοι τι ε, υποφέρουν. Όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την καλλιέργεια έχουν μεγάλο πρόβλημα. Κατά τρίτον, είπαμε ότι τα παιδιά δεν τρώνε αρκετά φρούτα και λαχανικά, άρα θα έπρεπε και η κυβέρνηση να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Οπότε θα πρέπει να μην υποτιμούμε το θέμα και δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε άκρα, οπότε το σχολείο να ομοκρατεί τους μαθητές σε σχέση με το τι τρώνε στο διάλειμμα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος, και τώρα ο κύριος Χόγκαν, ο Επίτροπος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μέλο για την έκθεσή του. Μου δίνει μια ευκαιρία για να εξετάσουμε κάποια από αυτά τα προβλήματα που έχουν σχέση με τον κλάδο των προγυπευτικών είπαμε για τη ρωσική απαγόρευση εισαγωγών και ισχύει και για τα προκυπτικά οπότε και πάλι βλέπουμε πόσο ευάλωτος είναι αυτός ο κλάδος. Γιατί έχουμε ε, αναταραχή στην αγορά, μια από αυτά τα προϊόντα είναι νομπού χαρακτήρα και αναλώνονται γρήγορα και θα πρέπει να κάνουμε για αυτούς τους ε, παραγωγούς. Καταλαβαίνουμε επίσης το πόσο βοηθάνε οι οργανώσεις των παραγωγών, πόσο κράτα πάνε σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Το Συμβούλιο είπε ότι θα πρέπει να ενδυναμωθεί η θέση τους σε σχέση με τους ε, μεγάλους λιανοπολιτές, ε, να βοηθήσουμε την καινοτομία, να έχουμε επίση κάποια μέτρα για πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων. Μπράβο στον κύριο Μέλλο, βοηθάει σε αυτή την προβληματική για το πώ μπορούμε να στηρίξουμε περισσότερο του οργανώσει παραγών, να είναι πιο αποτελεσματικέ ε, στα κράτη-μέλη και στα μέλλοντα κράτη-μέλη. Οπωσδήποτε, εμεί το θεματολόγιο μα, το πολιτικό, έχουμε προτεραιότητα αυτό το πρόβλημα, που το, το είπε και ο κύριο ε, Γιούνκερ, κάτι θα πρέπει να κάνουμε τον πρώτο δωδεκάμενο τη εντολή μα. Αυτό σημαίνει ότι θα καλύψουμε τα όσα αυτή η έκθεση, να βοηθήσουμε με ασφάλεια δικαίου και λιγότερο δικαιωτικό φόρτο τη οργανώση παραγωγών. Εμεί ε, φέτο πρόκειται να προβούμε σε απλούστευση των κανόνων ε, όσον αφορά την δική μας νομοθεσία. Οπότε έτσι θα είναι πιο ξεκαθαρό το νομικό καθεστώς. Δεν είναι κάποια μεταβολή φέτος. Αλλά θεωρούμε ότι είναι ακρογόνια η λίγη οργάνωση των παραγωγών και θα πρέπει να βοηθήσουμε αλλά δεν θα κάνουμε τώρα την, την αλλαγή ε, με πρωτογενή αλλά με δευτερογενή νομοθεσία αργότερα. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ βασικό το λειτουργεί αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων και εδώ θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αθέμητον αγωνισμό και αθέμητες πρακτικές. Πολλά κράτη-μέλη έχουν αρχίσει τώρα να κάνουν κάτι σε εθνικό επίπεδο. Η Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία ιδίω. Βεβαίω ο Γιώργος Κάλσκι Κύριε Μπιελκόφσκι είναι ο αρμόδιος επίτροπος, κυρία Μπιελκόφσκι, συγγνώμη, και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό για τις αθέμητες πρακτικές, για την αλυσίδα των τροφίμων και οι εκπρόσωποι είπαν ότι θα πρέπει να γίνει ανταλλαγή των πρακτικών ε, μια προσπάθεια το 2011 να έχουμε ένα ε, καθεστώς ε, το οποίο ισχύει σε ακούσια βάση το 2013 για την ε, αλυσίδα του εφοδιασμού. Επίσης είπαμε να νομοθετήσουμε για τις αθέμητες πρακτικές μέχρι το τέλος του εναστότος έτους. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία σας. Μπράβο στον κύριο Μέλο που μας βοηθάει για να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση του κλάδου των προκυπευτικών. Ευχαριστώ εδώ πέρα ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση και θα